Ε, βλέπουμε ένα νέο άνεμο να πνέει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με διάλογο πώς μπορεί η ΕΚΤ να σταματήσει τη χρηματοδότηση ρηπογόνων δραστηριοτήτων, πώς μπορεί να ε, προωθήσει την ισότητα των φύλων μεταξύ των ηθινόντων που παίρνουν τις αποφάσεις. Κάθε νέα θέση εργασία και δουλειά ξεκινάει με την πίστοση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει εκεί να γίνει πρόοδος, κυρία Λαγκάρτ, πραγματική. Η ΕΚΤ θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ε, βοηθήσει να εφαρμοστεί η ταξινόμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χρηματοδοτούνται ε, αποτελεσματικές και ουσιαστικές δράσεις. Και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στη βιωσιμότητα, τώρα που είναι χαμηλά τα επιτόκια, για να επανέλθει το πλήρες δυναμικό της νομισματικής πολιτικής. Εκεί συνεχίστε με εμπιστοσύνη σε αυτό το δρόμο και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ξαναβρούμε το σωστό δρόμο και εμείς και οι κεντρικές τράπεζες. Η κυρία Ανιές Βγέν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του 2018 που θα ψηφίσουμε αύριο στην Ολομέλεια θα είναι η πρώτη έκθεση, το πρώτο κείμενο που θα σας διαβάσουμε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω οι συστάσεις αυτές να επιτρέψουν και να αποτελέσουν τη βάση για να έχουμε τακτικό διάλογο με την Επιτροπή μας ΕΚΟΝ, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Σε αυτή την έκθεση βλέπετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας και η ΕΚΤ τα επόμενα χρόνια. Το Γενάρη στον Ταβός αναφερθήκατε στην ανάγκη να ενισχυθεί η αντίσταση ε, στο κυβερνοχώρο για τις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης εμβέλειας που θα επηρέαζαν σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία σε περίπτωση που γίνουν. Είναι κατεπήγον λοιπόν να ανακαινιστεί η αρχιτεκτονική της διεθνούς ευρωπαϊκής συνεργασίας. Να έχουμε κοινέ στρατηγικές και κοινέ προσπάθειες συντονισμένες για να αντιμετωπίσουμε τη ε, ψηφιακή μετάβαση. Υπάρχει ένα ρίσκο το οποίο πρώτα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το δεύτερο είναι να το αντιμετωπίσουμε με δράση. Ε, να είναι σε θέση να αντισταθούν τα συστήματά μας και να δούμε πώς συνεργάζονται οι τράπεζες της Ευρωζώνης. Ξέρω ότι μπορώ να ε, υπολογίζω στο δικό σας σθένο, αλλά, σθένος, αλλά και τη δέσμευση και την προσήλωσή σας προς την κατεύθυνση αυτή για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω 14 συναδέλφους. Θα πάρω εννέα. Ο κύριος Κίρτσος, παρακαλώ, από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαυρίδη για την πολύ καλή έκθεσή του και όσοι συνεργάστηκαν μαζί τους. Και να ευχηθώ στην κυρία Λαγκάρντ να έχει παρεμβάσεις εξαιρετικά σημαντικές που θα ακόμα πιο σημαντικές και από εκείνες του κυρίου Ντράγκη στην πορεία της ήθελα να, την, να προσθέσω δύο ερωτήσεις σε ένα βομβαρδισμό ερωτήσεων βέβαια. Η μία έχει σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή ξέρουμε ότι από το 2018 η κατάστασή του έχει γίνει καλύτερη αλλά θα ήθελα μία, αν μπορεί συνοπτικά να μας πει δύο πράγματα, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και πόσο γρήγορα. Και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος, τέθηκε από προηγούμενους συναδέλφους, είναι φανερό ότι για να πάμε στην πράσινη μετάβαση χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε πρόσθετες επενδύσεις και όπως έλεγε ο Ντράγκη και το 2018 αλλά και γενικότερα πρέπει να βελτιώσουμε τη σύνθεση των δημοσίων δαπανών ώστε να τις κάνουμε περισσότερο ποιοτικές και αν είναι δυνατόν επενδυτικές. Θα ήθελα λοιπόν κάποιο σχόλιο και από την κυρία Λαγκάρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρκες. Μάρκες. Μάρκες Η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Μαυρίδη, να σα ευχαριστήσω για την εκθεσή σα. Κύριε Λαργάρντα, σα ευχαριστούμε για την παρέμβασή σα. Προφανώ θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Μέχρι στιγμή η πρόοδο αφού ήταν πολύ αργή και περιορισμένη. Ο τρίτο πυλώνα τη Τραπεζική Ένωση ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω ότι αν θέλουμε ένα ισχυρό ευρώ θα πρέπει καταρχάς να έχουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση πίσω από το ευρώ, στο πλευρό του νομίσματος αυτού. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα δημοσιονομικό εργαλείο το οποίο θα μπορεί να αντέχει τελικά σε εξωτερικούς κλειδονισμούς και για τα 27 κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν μπορεί να δραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο και μπορεί καθοριστικό ρόλο επίσης να, αντιδραματίσει και στην επεντόπιση κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και με εξωτερικούς και διεθνείς φορείς προκειμένου το ευρώ να γίνει ισχυρό αποθεματικό νόμισμα ιδίω στους διεθνείς οργανισμούς όπου έχει παρουσία το νόμισμα αυτό. Πέκαρινεν. Ο κύριος Κέρελα. Uh, uh, Ευχαριστώ. Να πω εξ αρχή, κυρία Λαγκάρδο, ότι θέλω να θέσω το ζήτημα του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και τι επιπτώσει αυτού στι ευρωπαϊκέ οικονομίε όσον αφορά τη δυνατότητα επενδύσεων στην, στο πλαίσιο τη Πράσινη συμβασία, αλλά και για τα κίνητρα που δίνονται, τα κανονικά, τα παραδοσιακά ε, δημοσιονομικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, νομίζω ότι η Κομισιόν εκτελεί μια ε, αξιολόγηση το επόμενο διάστημα αυτού του Συμφώνου. Και θα ήθελα να μάθω αν η ΕΚΤ πρόκειται να αποκτήσει έναν ε, επίσημο ρόλο όσον αφορά την παρακολούθηση αυτού του συμφώνου και αν θα τροφοδοτήσει τι σχετικέ συζητήσει. Γιατί αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία, πιστεύω ότι το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη είναι υπερβολικά περιοριστικό όσον αφορά τη δυνατότητα κυβερνήσεων να επενδύουν σε οικονομικά στοιχεία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και τέλο, θα ήθελα να εξετάσετε και τις Ιρλανδικές τράπεζες και τα επιτόκια που χρεώνουν για δάνεια και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας υπόψη ότι στην Ευρωζώνη, σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, οι δικές μας τράπεζες δίνουν δύο, χρεώνουν δύο και τρεις φορές τα, ε, ε, τα επιτόκια που δίνουν άλλες τράπεζες στην Ευρώπη, ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια και ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Φερέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως υπόθηκε και πριν από λίγο, οι πολιτικές συνομισματικές που ακολουθήθηκαν πραγματικά δεν αρκούσαν τελικά για να αντιμετωπίσουμε την δινή οικονομική κατάσταση την οποία γνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πρόβλημα είναι ότι ενδεχομένως να πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μια επερχόμενη οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση τα συμβατικά μέτρα είναι αρκετά περιορισμένα. Συνεπώς λοιπόν θα φανούν ε, ότι ορισμένες χώρες τελικά αυτές που είναι στην Ευρωζώνη θα είναι ακόμα πιο ευάλωτες στο μέλλον. Πολλές φορές έχουμε δημοσιονομική πολιτική η οποία αντιβαίνει στους καλούς μισθούς ή επενδύσεις, δεν προωθεί τις δημόσιες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δημοσιονομική πολιτική η οποία να είναι θετική για την οικονομική ανάπτυξη και η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Ακριβώ όμω εδώ έγκυται η παγίδα, η παγίδα του ευρώ. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψουμε το ευρώ το στομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ο κ. Καστάλτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο δρόμος προς μία πιο ισχυρή οικονομική και νομισματική ένωση ακόμα βρήθη ερωτήσεων στις οποίες δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Πρέπει να βρεθούν λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Πολύ αργή και μόνο ήταν η πρόοδος που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ορισμένα προγράμματα και σχέδια αρκετά αμφιλεγόμενα τελικά εφαρμόστηκαν. Η βασική όμως πρόταση για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης τελικά από ό,τι βλέπουμε δεν σημειώνει επαρκή πρόοδο καθότι η Ευρωζώνη εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, ιδίω όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης των Καταθέσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει καταθέσει των Ευρωπαίων πολιτών. Μέσω όμω του ΕΔΙΣ, του Ευρωπαϊκού Αυτού Συστήματο, θα καταφέρναμε τελικά να προασπίσουμε τι καταθέσει αυτέ και μάλιστα να δημιουργήσουμε πιο ισχυρά οικονομικά συστήματα που θα ήταν πιο ανθεκτικά στι οικονομικέ κρίσει. Δεν νομίζω πάντω ότι μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μόνο στο κριτήριο του κινδύνου, του ρίσκου, προκειμένου να δημιουργήσουμε το Ευρωπαϊκό Αυτό Σύστημα Ασφάλιση Καταθέσεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, είναι παράλογο. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα έχουμε ένα οικονομικό ευρωπαϊκό σύστημα ακόμα πιο ασθενέ. Νομίζω ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να λάβουμε δράση, διαφορετικά το τίμα θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, χαίρομαι που σα βλέπω εδώ, κυρία Λαγκάρτ, μετά το διορισμό σας. Και θα πρέπει να συγχαρούμε τον προκάτοχό σας, τον κύριο Ντράγκη, που κράτησε σταθερό το ευρώ και την ευρωζώνη και την ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να σας δώσω το εξή. Είχαμε εκλογές στην Ιρλανδία και κυριάρχησε το θέμα της στέγασης. Αναφέρθηκε ο κύριος Κελεχέρ στα επιτόκια. Δεν είναι μόνο τα επιτόκια, είναι και οι κανόνες δανεισμού. Και έχουμε τώρα μια κατάσταση όπου ο κόσμος έχει υψηλή μόρφωση, πάρα πολύ καλές δουλειές και δεν έχει λεφτά να πάρει σπίτι. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο για την προσφορά που δεν είναι μεγάλη, αλλά ακόμα και όταν υπάρχει προσφορά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και πολλοί κόσμος τώρα μένει με τους γονείς του ακόμα γιατί δεν μπορεί να δανειστεί να αγοράσει σπίτι. Σας λέω άνθρωποι με καλή εκπαίδευση, με καλές δουλειές που καλοπληρώνονται αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι λόγω των κανόνων που ισχύουν και εφαρμόζουν οι τράπεζες για τις χορηγήσεις. Μπορείτε λίγο να χαλαρώσετε εκεί τα πράγματα για να δώσετε λίγη ελπίδα στους ανθρώπους αυτούς. Για να ξέρουν ότι αυτό που μπορούσες να έχεις στο παρελθόν, μια καλή δουλειά και ένα καλό σπίτι, θα συνεχιστεί. Ο κύριος Ρουίθ Τεβέσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Λαγκάρτ. Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης. Καταρχάς θα ήθελα να διαβιβάσω την υποστήριξή μου στην έκθεση του συναδέλφου Κώστα Μαυρίδη της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Είναι πάρα πολύ πλήρης η έκθεση αυτή και περιλαμβάνει πολύ ουσιαστικά στοιχεία. Κάτι πρόσθετο ενδεχομένως και στη γραμμή των όσων είπε ο κύριος Φερνάντεθ, ο σοσιαλιστής ε, εκπρόσωπος είναι τα νέα μέσα και τα νέα ε, εργαλεία. Δεν είναι μόνο τα πολύ χαμηλά επιτόκια και αγορά ε, ομολόγων που θα φτάσει ε, στο στόχο. Χρειάζεται και υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει όμως άνευ όρων να υποστηρίζει τους στόχους. Θα υπάρξουν άμεσες ε, μεταφορές πιστώσεων προς τα νοικοκυριά των όσων ζουν στην Ευρωζώνη για να τονωθεί η κατανάλωση. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώθηκε εδώ η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΕ. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Ντομπρόφσκης, να πάρει το λόγο για να κλείσει η συζήτηση. Κύριος Ντομπρόφσκης, παρακαλώ. Mr. Chair, Madam President. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, έδειξε η συζήτηση ότι υπάρχει ε, σύγκληση απόψεων όσον αφορά τις περισσότερε διαστάσεις τη έκθεσης και χαίρομαι που βλέπω αυτό το κοινό έδαφο που ε, φαίνεται να ε, υπάρχει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Θέλω να αναφερθώ στα ζητήματα που απευθύνθηκαν στην Κομισιόν. Ε, ζητήθηκε από την Κομισιόν να εξετάσει ε, ζητήματα όπως το ψηφιακό νόμισμα της ΕΚΤ. Όπως ε, πολλές ε, κεντρικές τράπεζες, η Κομισιόν και η ΕΚΤ πλέον ε, αναλύουν πιθανά ωφέλη αλλά και πιθανούς κινδύνους όσον αφορά αυτά τα νομίσματα. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αλλά δείχνει τουλάχιστον η διαδικασία αυτή ότι τα τρία θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου μπορούν να αλληλεπιδρούν όσον αφορά βεβαίω εντό των αρμοδιοτήτων του ο καθένα. Οπότε περιμένουμε τη δική σα υποστήριξη για να ενισχύσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Πρόεδρε. Να καλέσω τώρα την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κυρία Λαγκάρτ, να λάβει το λόγο και να την ευχαριστήσω ε, για την πολύ ευγενική και φιλική δεξίωση που διοργανώθηκε χθες στην Γαλλία στην, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κυρία Λαγκάρτ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου. Α, ναι, έπρεπε να σηκωθώ για να μιλήσω. Ναι, δεν το ήξερα, ζητώ συγγνώμη. Ε, δεν ήξερα ότι έπρεπε να σηκωθώ για να μιλήσω όρθια στο ε, Κοινοβούλιο Θα προσαρμοστώ και θα συμμορφωθώ στους κανόνες. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το διάλογο αυτό που είχαμε και αποτελεί πραγματικά τμήμα των όσων εμείς θεωρούμε στην ΕΚΤ και στο Ευρωσύστημα ως απαραίτητο για να έχουμε διάλογο με την κοινή γνώμη, με την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους της, αλλά κυρίως εκείνους που εκπροσωπούν τους πολίτες της Ευρώπης, εσάς δηλαδή, τα μέλη του Κοινοβουλίου που έχετε εκλεγεί από τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό πραγματικά αποτελεί τμήμα της λογοδοσίας που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και προς εσάς αλλά και προς τους πολίτες της Ευρώπης μέσω ημών. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές τους τελευταίους μήνες και μία από αυτές που θέλω οπωσδήποτε να εφαρμοστεί όσο προχωρούμε στην ε, στρατηγική αναθεώρηση είναι ο μόνιμος διάλογος που θέλουμε να έχουμε. Αυτό που ονομάζουμε ε, outreach, ε, δηλαδή ε, απευθυνόμαστε σε εσά και στους πολίτες της Ευρώπης. Να σας αναφέρω μερικά σημεία για την αναθεώρηση στρατηγική μας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ορισμένοι από εσά μιλήσατε για την νομισματική πολιτική και τα σημερινά στοιχεία που χρησιμοποιούμε για να εφαρμόζουμε την πολιτική μας από το 2014 και εντεύθεν. Για ε, όσους λέγουν ότι αυτή εδώ η νομισματική πολιτική και ιδιαίτερα τα μη συμβατικά εργαλεία ήταν αντιπαραγωγικά, θέλω να απαντήσω στεναρά και να τους πω κοιτάξτε τον αντίκτυπο αυτών των αντισυμβατικών μέτρων και εργαλείων. Πώς επηρέασαν την οικονομία, πώς αυξήθηκε η ανάπτυξη και πώς οι οικονομίες μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη κυρίως είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από ό,τι θα βρισκόντουσαν αν δεν χρησιμοποιούσαμε αυτή την αντισυμβατική πολιτική. Βεβαίως όλα αυτά μπορούν να μετρηθούν με ποσοτικούς όρους. Δεν εννοώ αυτό όμως. Μπορεί να είναι 2,5 με 3% περιφερειακή ή περιθωριακή η αύξηση. Ταυτόχρονα όμως ε, έχει ε, συνεισφέρει η πολιτική μας και για τον πληθωρισμό. Και ξέρετε ότι το 2003 αναθεωρήθηκε η στρατηγική. Ε, έχουμε μετρήσεις και σε σχέση με τον πληθωρισμό. Αυτά τα αντισυμβατικά εργαλεία λοιπόν που χρησιμοποιήθηκαν από το 2014 βοήθησαν για τον πληθωρισμό για να αυξηθεί λίγο. Ε, θα θέλαμε να είναι και λίγο παραπάνω σε συνδυασμό με άλλα μέτρα. Περίπου μισή ποσοστία μονάδα αυξήθηκε ο πληθωρισμός, που σίγουρα δεν είναι κακό δεδομένο το επίπεδο ε, στο οποίο βρισκόμαστε. Κάποιοι μιλήσατε για πληθωρισμό 1%. Ήταν 1,3% το οποίο σίγουρα δεν είναι ο στόχος μας, αλλά παραπάνω από το 1% που ακούστηκε. Αυτά λοιπόν τα μη συμβατικά μέτρα και εργαλεία που χρησιμοποίησαμε βοήθησαν τις οικονομίες μας και εξακολουθούν και σήμερα να το κάνουν. Αν κοιτάξετε απλώς τον όγκο και τον αριθμό των νέων χρηματοδοτήσεων στην πραγματική οικονομία, είτε είναι στις επιχειρήσεις είτε στα νοικοκυριά, βλέπουμε μια χρηματοδότηση που είναι πολύ χαμηλή σε κόστος και σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε για τις Ιρλανδικές τράπεζες και πόσο χρεώνουν και ποια επιτόκια επιβάλλουν και το κοιτάμε αυτό οπωσδήποτε. Αλλά το κόστος του δανεισμού ε, είναι χαμηλότερο για την πραγματική οικονομία, ένα αυτό. Και δεύτερον, οι ε, χρηματοδοτήσει τη οικονομία αυξηθήκανε και εξακολουθούν να αυξάνονται. Μπορεί να είδατε κάποια σχόλια πρόσφατα ότι ε, συνεχίζεται αυτό και αυξάνεται βέβαια λιγότερο για τα νοικοκυριά και περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Είναι γεγονός. Γενικά πάντως ήταν πολύ θετική επίπτωση για τις οικονομίες μας. Και ως τμήμα της αναθεώρησης στρατηγικής μας είναι ακριβώς να αξιολογήσουμε και ποσοτικά και ποιοτικά αυτή την εξέλιξη και ιδιαίτερα να κοιτάξουμε τις παρενέργειες και ενδεχομένως τις ισορρευμένες, ισορρευτικές παρενέργειες που θα μπορούσε να έχει στους πολίτες και στις οικονομίες. Τώρα, ένα δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω σύντομα, επικεντρώθηκα στη νομισματική πολιτική και τα μέσα και τα εργαλεία και πώς τα μετράμε και πώς τα κοιτάμε και ε, τα ωφέλη όχι μόνο τα αρνητικά είναι κλιματική αλλαγή. Ουδής μπορεί να ζητάει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να υποκαταστήσει τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Ως πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι ένα από τα βασικά εργαλεία για την κλιματική αλλαγή είναι η τιμολόγηση της ενέργειας. του άνθρακα. Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει καμία κεντρική τράπεζα να το αποφασίσει. Και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις πολιτικές μας. Και τη σταθερότητα των τιμών, που είναι ο πρώτος στόχος, και πώς επηρεάζει αυτόν τον στόχο. Ή σε σχέση ακόμα και με τη διαχείριση του κινδύνου. Γιατί εμείς είμαστε υπόλογοι και σε εσά και στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, αν δείτε τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων που διαχειριζόμαστε και πού είναι το ρίσκο και πώς συνδέεται το ρίσκο της κλιματικής αλλαγής με κάποιες εγγυήσεις που έχουμε στα χαρτοφυλάκια μας και αν αυτό ε, μετράμε ή όχι. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν θα είναι από τα θέματα που θα λάβουμε υπόψη μαζί με τα πιο παραδοσιακά στοιχεία που θα μετρούμε. Στα πλαίσια αυτή τη αναθεώρηση λοιπόν τη στρατηγική μα, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο όχι μόνο μαζί σα, αλλά και με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, Προηγουμένω ήταν εδώ η πρόεδρο τη Επιτροπή και πολλά μέλη τη Επιτροπή παρίστανται. Θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το διάλογο και πραγματικά θέλουμε να είναι διπλή κατεύθυνση αυτό ο δρόμο, όχι μονόδρομο. Ευχαριστώ για τι ειδικέ ερωτήσει για τι χώρε. Ε, να το δούμε διμερώς, δεν θα ήθελα να απαντήσω εδώ σε αυτό. Ε, αν σας ενδιαφέρουν οι ειδικέ τράπεζες ή κάποιες χώρες συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προσωπικά και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των γενικών συμφερόντων της, θέλουμε να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Λοιπόν, ο Κώστας Μαυρίδης έχει τον λόγο ε, ο εισηγητής για αυτό το σημείο της σημερινής σας διάταξης. Παρακαλώ. Thank you, Mr. I be short too. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Δύο σημεία θέλω να θίξω. Κυρία Λαγκάρντα, σήμερα είδατε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να έχουμε αποκλίνουσες απόψεις. Σκεφτείτε λίγο το παρελθόν. Σκεφτείτε λίγο τη στάση του κυρίου Ντράγκη. Ο κύριο Ντράκη μπορεί να μην υπήρξε τελικά τέλειο, αλλά η παρακαταθήκη του τελικά είναι ότι ήταν αποφασισμένο να σώσει την Ευρωζώνη. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ενδεχομένω να έσωσε ακόμα και το ευρωπαϊκό όραμα, το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και ορισμένοι μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να το συγχωρήσουν γι' αυτό. Μα είπατε πολύ σωστά σήμερα στην αρχική σα παρέμβαση ότι ε, ουσιαστικά μοιραζόμαστε την ίδια άποψη όσον αφορά τι προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα πρόστα και κάτι ακόμα. Ακόμα και ο κύριο Ντομπρόμφσκης και εν γέννη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν την ίδια άποψη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρόσθετα ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, όπως αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, λείπουν εδώ πέρα. Νομίζω ότι η βασική πρόκληση για όλους είναι να καταφέρουμε να έχουμε συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα για τον Ευρωπαίο πολίτη και για να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών με πολλού συγκεκριμένου τρόπου. Ολοκλήρωση Τραπεζική Ένωση, ολοκλήρωση τη Ένωση Κεφαλαγορών και πολλά άλλα πράγματα. Συνεπώ, εναπόκειται σε εσά, κυρία Λαγκάρντ, και θα σταθούμε εμεί στο πλάι σα να καταφέρουμε να έχουμε μια πραγματική σύγκληση των ευρωπαϊκών οικονομιών. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά. Και με αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την παραβίαση της απόφασης 2017-2074 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα. Παράνομη είσοδο στην επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσώπη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κυρώσεων. Θέλω λοιπόν να καλέσω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μπορέλ, να τον καλωσορίσω καταρχάς. Κύριε Μπορέλ, είστε έτοιμος. Ο κύριος Μπορέλ βρίσκεται εδώ με την ιδιότητά του ως είπα το εκπροσώπου του εκ μέρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα συζήτηση σήμερα αφορά μια εικαζόμενη ε, παραβίαση περιοριστικών μέτρων στη Βενεζουέλα. Η σχετική απόφαση λήφθη το 2017 ως, προσπα... ως μέρος των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης ε, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα. Αυτό το, αυτή η απόφαση ε, ε, περιλάμβανε και την απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και 25 ατόμων μεταξύ αυτών και της Ντέλση Ροντρίγες που ήταν αντιπρόεδρος ε, της ε, Βενεζουέλας. Αυτή η απόφαση καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτραπεί η είσοδος ή η διέλευση των ε, ατόμων αυτών από την επικράτειά της. Γνωρίζετε ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα σε όλες τις περιπτώσεις για την εφαρμογή και την επαλήθευση ε, κυρώσεων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική τους ένωμη τάξη. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα, επαναλαμβάνω, σε όλες τις περιπτώσεις για την ε, εφαρμογή και την επαλήθευση των κυρώσεων που έχουν ε, εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο, όταν μια πιθανή παραβίαση αυτών των κυρώσεων ανακύπτει, για παράδειγμα κάτι που σχετίζεται με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων ή απαγόρευση εισόδου, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που πρέπει να ερευνήσουν και να καθορίσουν αν πράγματι έχει υπάρξει μια τέτοια παραβίαση. Όσον αφορά την ευρύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των κυρώσεων, η Κομισιόν έχει εποπτικό ρόλο όσον αφορά τον ομοιόμορφο τρόπο εφαρμογής αυτών των κυρώσεων ε, με βάση πάντοτε τις αρμοδιότητές της. Αυτό, για παράδειγμα, ισχύει με το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και κάποιους, κάποια κλαδικά ζητήματα, αλλά αυτό δεν αφορά απαγόρευση εισόδου. Μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίω την καταλληλότητα από πολιτική άποψη τα κράτη-μέλη να ε, εκχωρήσουν αυτή την αρμοδιότητά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω κάτι τέτοιο βεβαίω θα απαιτούσε ε, τροποποίηση τη συνθήκη. Όμω Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και σαφής. Η Κομισιόν δεν μπορεί με δική της πρωτοβουλία να ξεκινήσει η διαδικασία επιπαραβάση όσον αφορά πιθανή ε, παραβίαση απαγόρευσης εισόδου στην επικράτειά της. Αυτές οι απαγορεύσεις εισόδου περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου και γι' αυτό δεν εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Κατά τη συνέπεια, η Κομισιόν δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο όσον αφορά την παρακολούθηση τη εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, ούτε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Ω ύπατο εκπρόσωπο που βρίσκομαι εδώ και ω εκπρόσωπο του Συμβουλίου, είμαι υπεύθυνο επίση για να εξασφαλίσω ε, την ε, ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ε, άμυνας συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που έχουν εγκριθεί σε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου είμαστε αρμόδιοι. Ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, βεβαίω, πάντοτε βρισκόμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν εικαζόμενε παραβιάσει, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι οι κυρώσει που έχουν εγκριθεί θα επιβάλλονται με ομοιογενή, ομοιόμορφο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Μπορέλ. Ερχόμαστε στη συζήτηση τώρα. Κυρία Μονσεράτ, πρώτη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Βενεζουέλα και η πολιτική της Βενεζουέλας έφτασαν στην Ισπανία ε, από το χέρι του Ιγκλέσιας και του Μονεδέρο. Δεν τα είπα εγώ αυτά. Ο Πέδρο Σάντσεθ, που είναι τώρα πρωθυπουργό στην Ισπανία το 2016. Και τώρα γνωρίζουμε ότι δεν ήταν κριτική αυτό για εκείνον, αλλά ήταν έπαινος. Σήμερα ο Ιγκλέσιας είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και η πολιτική του Τσάβες λερώνει την εικόνα της κυβέρνησης η κυβέρνηση Σάντσεφ ε, άνοιξε τις πόρτες στον τσαφισμό. Ο Άμπαλος, ο υπουργός ε, ε, σοσιαλιστής, σε συνάντησε την Τέλση Ροντρίγκες, αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, του Μαδούρο, της δικτατορίας σε ευρωπαϊκό ε, έδαφος και παραβιάζει έτσι ε, τις αποφάσεις και τις κυρώσεις και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, η κυβέρνηση Σάντσεθ ψεύδεται και δεν ε, εφαρμόζει τα συμφωνηδέντα. Έχει χάσει κάθε αξιοπιστία και θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να διερευνήσουν την αλήθεια. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι αδελφός του ισπανικού λαού. Έχουμε εκατομμύρια Βενεζολάνους, τους οποίους καταπατά ο τύρανος Μαδούρο και για αυτού και για εκείνου που έχουν έρθει στη χώρα μας θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, να γίνεται σεβαστό το καθεστώ των κυρώσεων. Για μας τους Ισπανούς και τους Ευρωπαίους και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα είμαστε υπέρ της ε, ελευθερία στη Βενεζουέλα. Να ψάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έγινε, να βρεθεί αλήθεια και να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο σκάνδαλο το οποίο ντροπιάζει την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μονσεράτ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος Μορένο Σάντσεφ. Κυρία Μονσεράτ, έχετε μια ερώτηση με μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Μονσεράτ αν θεωρεί σκόπιμο να χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εργαλείο για να επιτεθεί στην Ισπανική κυβέρνηση, λέει η κυρία Μέστρε. Γνωρίζοντα ότι το κοινοβούλιο μα εδώ δεν έχει τέτοιε αρμοδιότητε. Αν το θεωρείτε σκόπιμο, μήπω έρθουν και άλλε πολιτικέ ομάδε να φέρουν ε, θέματα εθνικού ενδιαφέροντο που ενδιαφέρουν πολλού στην Ισπανία. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά δύο πρωθυπουργοί πρώην, ο Αθνάρ και ο Ραχώη. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Σας επισημαίνω ότι στη γαλάζια κάρτα έχουμε 30 δευτερόλεπτα ε, για την ερώτηση και για την απάντηση και χωρίς προειδοποίηση με το σφυράκι θα σας ε, κόψω. Τι είναι αυτά τα στάχτες στα μάτια. Εσείς κάνετε εκστρατεία κατά της Ισπανίας. Ανοίγετε τις πύλες της Ευρώπης στον τσαβισμό. Εσείς τα ξέρετε, παραβιάσατε τις κυρώσεις και ψεύδεστε. Εξηγήστε γιατί. Εσείς έχετε χάσει όλη την αξιοπιστία και θέλετε να τη χάσουμε και όλοι οι Ισπανοί μετά από εσά. Γι' αυτό σας ζητούμε να πάρετε εσείς τις αποστάσεις σας από το λαϊκισμό και τον τσαβισμό προσαρτηθείτε και πάλι εδώ και τώρα στο άρμα της Ευρώπης. τώρα ο συνάδελφος Μορένο Σάντσεθ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Ντολόρες, Τζόμπι, 9 από τους 10 ομιλητές είμαστε Ισπανοί σε αυτή τη συζήτηση και ρωτώ σε όσους έφεραν την ε, πρωτοβουλία αυτή. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι ευρωπαϊκή αυτή η συζήτηση. Μήπως γελιοποιούμαστε εδώ θα συνεχίσετε να εκμεταλλεύεστε το Κοινοβούλιο για να κάνετε αθέμητη αντιπολίτευση ε, στην ε, Ισπανία. Ε, κύριοι του ΕΛΚ, των Θιουδαδάνος και του Βόξ, εσείς πλήτετε σφοδρά την εικόνα της Ισπανίας εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο. Ούτε ένα λεπτό δεν σκεφτήκατε το λαό της Βενεζουέλας που αυτό που περιμένει από εμά είναι στήριξη και ενότητα και όχι διχασμό και σύγκρουση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας δρά και έδραση ε, ω συνομιλητή αναγνωρισμένο από συμπολίτευση και αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα για μια ε, πορεία προ δίκαιε και ελεύθερε εκλογέ ω έντιμο διαμεσολαβητή. Και τότε το Κοινοβούλιο θα στείλει επιτροπή αποστολή παρατήρηση εκλογών. Σα παρακαλώ λοιπόν, μάθετε να δουλεύετε εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο και μην γελιοποιήστε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γόλας. Κύριε Μορένο Σάντσεφ, ε, δέχεστε ερώτηση του κυρίου ε, Γόλας, του συναδέλφου. Πείτε. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο τελευταίος ομιλητής μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, αναγνωρίζοντας εδώ πέρα τη θέση Ισπανίας. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ε, έχουμε δει τη στάση Ισπανίας σε πάρα πολλές πτυχές της πολιτικής της Βενεζουέλας. Δεν θεωρείτε ότι η αναγνώριση του Γκουάιδο αποτελεί πραγματικά επονίδιστη στάση για οποιονδήποτε βρίσκεται εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί πραγματικά μία επέσχυντη στάση για πάρα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Μαρένο Νομίζω ότι το είπα προηγουμένως. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας είναι συνεπής. Αυτό που θέλουμε είναι να ζητήσουμε μια λύση με όλους τους Βενεζουελάνους. Η διαφορά είναι ότι εμείς επιζητούμε το διάλογο και όχι τη σύγκρουση και το διχασμό. Λύση θα βρεθεί μόνο έτσι. Γιατί ε, υποφέρει ο λαός της Βενεζουέλα. Θα πρέπει να τους ενώσουμε εμείς, όχι να τους διχάσουμε. γι' αυτό η Ισπανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να βρει μια λύση, όπως σας είπα, με διαπραγμάτευση, με δημοκρατία, με συνεννόηση και ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Κύριε Γόλας. Ε, σας ε, επιπλήττω για μια έκφραση που χρησιμοποιήσατε. Ε, ο κύριος Κάνιας έχει το λόγο. Ε, Τώρα θα προσπαθήσω να ξεπεράσω αυτή τη λάσπη των σοσιαλιστών, αλλά θα τα καταφέρω. Κύριε Μπορέλ, εγώ θα ήθελα να σας ακούσω να μιλάτε ως ύπατος εκπρόσωπος και όχι ως πρώην Υπουργός Εξωτερικών του κυρίου Σάντσεφ. Και να σας πω γιατί αυτή δεν είναι συζήτηση εθνική, είναι μια συζήτηση για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και σεβασμού στο Κοινοβούλιο. Πώς σέβεστε το κοινοβούλιο με αυτές εδώ πέρα τις φιλιαρίες. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Σεβασμός εδώ τι σημαίνει. Ε, ζητήσαμε να ενταθούν οι κυρώσει κατά του Μαδούρο και του καθεστώτος με τις δικές σας ψήφους. Και όταν μια κυβέρνηση αποφασίζει να ε, παραβιάσει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, τότε αυτό είναι εις βάρος της αξιοπιστίας μας και όλων των θεσμικών οργάνων. Οι υπόλοιποι πώς να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα ίδια της τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τις αποφάσεις που παίρνει το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα. Θυμίζω ότι Αυτά τα ψηφίσματα και αποφάσεις δεσμεύουν τους πάντες και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η Επιτροπή είναι θεματοφύλακας όλων αυτών και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας δεν ήταν ειλικρινή. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδράνησε. οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε κάποια έγγραφα εξαίρεση του κυρίου Μαδούρο. Έχετε κοινοποιήσει τίποτα. Δεκάρα δεν δίνεται για όλα αυτά. Δεν έχετε το λόγο κύριε Σάντσεθ. Ε, ούτε ε, εσείς κύριε Κάνιας. Κοιτάξτε. όταν έχω κόψει το λόγο από συνάδελφο που έχει μακρηγορήσει μετά από 30 δεύτερα δεν θα του ξαναδώσω μπλε κάρτα, έτσι ήθιστε. Ο κύριος Ουρτάσουν Μα δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα, γιατί η απόφαση και οι κυρώσει του Συμβουλίου είναι εθνική αρμοδιότητα. Εδώ φέρανε μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει στην Ισπανική Βουλή. Και θέλω να στήσω συγγνώμη από όλου του συναδέλφου που απασχολούμε τώρα τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα εθνικό θέμα. Ε, εννιά Ισπανοί είναι ομιλητέ για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνετε, είναι αξιοθρύνητη η κατάσταση. Επιπλέον, θέλω πάρα πολύ ειλικρινά να πω ότι για τέτοια πράγματα όταν τα κάνουμε έτσι υποβαθμίζουμε και την ίδια την εικόνα της ισπανικής αντιπροσωπείας των Ισπανών Ευρωβουλευτών εδώ μέσα. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια και θέλω να πω κάτι στους ευρωπαϊκούς συναδέλφους του ΕΛΚ. Τη Δευτέρα ψήφισαν να γίνει αυτή η συζήτηση και σήμερα απουσιάζουν. Κάθε φορά που θα έχουμε μια συζήτηση εσωτερικής πολιτικής θα το φέρνουμε εδώ και τι θα το καταντήσουμε εδώ πέρα το κοινοβούλιο. Θέλω λίγο σεβασμό και λίγη ευθύνη γιατί έχουμε πολλέ δουλειέ και πάρα πολλέ σοβαρέ να ασχοληθούμε αντί να συζητάμε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξαναπώ, επειδή τέθηκε το ερώτημα. Εγώ προσωπικό, προσωπικά πάντοτε όταν κάποιος, όταν έχω αφαιρέσει το λόγο από κάποιον επειδή έχει υπερβεί το χρόνο αγόρευσή του, τότε δεν θα τον επιβραβεύσω δίνοντάς του τη δυνατότητα μέσω μπλε κάρτας. Το ίδιο θα κάνω και στην περίπτωση του κυρίου Κάνιας. Ο κύριος Στέρτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Μπορέλ, εμείς στο Συμβούλιο, η Κομισιόν, ανακατευόμαστε παντού και τώρα έχετε το θράσος να μας λέτε ότι ανακατευόμαστε όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή απόφαση να επιβληθούν κυρώσεις σε μια σειρά από εγκληματίες αυτή τη μαφία την κομμουνιστική και ναρκολαθρέμπορη που κυβερνάνε. Πολύ θράσο έχετε που θα λέτε ότι είναι και παρέμβαση αυτά στα εσωτερικά, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν ασχολούμαστε με την εκπαίδευση στην Ουγγαρία, με τη δικαιοσύνη στην Πολωνία και δεν συμμαζεύεται. Και προ Θεού, μην λέμε ότι είναι εσωτερική συζήτηση τη Ισπανία. Είναι μια συζήτηση για το σεβασμό των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χονδροειδώ παραβιάζει μια σοσιαλκομμουνιστική κυβέρνηση που έχουμε τώρα εδώ και ένα μήνα στην Ισπανία και όπου ήδη έχει συναντηθεί παράνομα με ένα εγκληματικό καθεστώ σε Ισπανική επικράτεια. Ποιο ξέρει για ποιο λόγο, ποιο ξέρει με ποιε προποθέσει και για ποιο μυστηριώδη ε, κίνητρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τέρτς. Για ένα λεπτό η κυρία Βιλανοέβα Ρουίθ. Κοιτάξτε, είναι τελείως χονδροειδές και ε, ανεύθυνο να χειραγωγείτε για άλλη μια φορά το λαό της Βενεζουέλας. Αλλά σιγά μη σας νοιάζει τώρα ε, η Βενεζουέλα. Είναι μια χώρα διχασμένη που χρειάζεται ευθύνη, που χρειάζεται να σταματήσουμε τις κυρώσεις γιατί ο λαός υποφέρει. Θα γίνουν εκλογές και να γίνουν με εγγυήσεις. Είδαμε τον κύριο Τέρτς να στέλνει μήνυμα σε όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για μεγάλο άγχος και αγωνία για το ποιο συνάντησε ποιο υπουργό. Αγωνία ε, δημιουργείται στους νέους μας ε, στους γεωργούς που δεν παίρνουν ε, σωστές τιμές ή το ρεύμα που κόβεται στη Γρανάδα όπως είναι η Εντέσα, η ΔΕΗ της Ισπανίας, η πολυεθνική. Αλλά εσάς καρφάκι δεν σας καίγεται για τους πολίτες. Μόνο οι ελίτ σας νοιάζουν ε, να υποδαβλίζετε τις συγκρούσεις, τις ένοπλες σειράξεις. Η χώρα μας, η Ισπανία, είναι πολύ καλύτερη από το άσπρο μαύρο που θέλετε εσείς να ε, ζωγραφίσετε. Ε, ο κόσμος και ο λαός στην Ισπανία έχει μέλλον και όχι αυτό που θέλετε εσείς. Ευχαριστώ. Και εδώ δεν θα επιτρέψω μπλε κάρτα και τον λόγο δίνω στον συνάδελφο Λόπεθ Χίλ. Είναι γεγονό ότι εδώ δεν είναι μια συζήτηση για την Ισπανία ούτε για τη Βενεζουέλα. Είναι απαραίτητη η δράση μας για την αξία των κυρώσεων και για τις αρχές μας. Υπάρχουν κάποιες αρχές ενδογενείς και εγγενεί ε, για τη δημιουργία της Ένωσης. Το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια, την ε, νομιμότητα. Πρόσφατα μάθαμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση ε, γελιοποίησε τι κυρώσει που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018. Αυτά τα μέτρα απαγορεύουν την είσοδο σε ευρωπαϊκή επικράτεια στην αντιπρόεδρο του καθεστώτος Μαδούρο και κυρώσεις που τους ε, πλήττουν γιατί υβρίζουν την Εθνοσυνέλευση και καταπατούν την δημοκρατία. Το Συμβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει σε βάθος αυτό και ε, τις κυρώσεις και στο ρελέξ να ενημερωθεί ε, στη συνέχεια το Κοινοβούλιο αρμοδίως. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε ε, τα κράτη. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Λόπεθ Χίλ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η συνάδελφο Κονθάλεθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γεγονό. Τούτη εδώ η συζήτηση δεν είναι ευρωπαϊκή. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει στην Ισπανική Βουλή. Γελιοποιήστε και δεν πάνε να κάθεστε όλοι εκεί μαζί. Μειοψηφία είστε και ούτε στην Ισπανική Βουλή έχετε πλειοψηφία. Ζητώ συγγνώμη από του υπόλοιπου βουλευτέ που θα πρέπει να ανεχθούν τώρα μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει στην Ισπανική Βουλή. Η, ε, η δική σα πολιτική δύναμη θα χαθεί. Δεν έχετε παρά δέκα βουλευτές. Ε, ε, είστε ασήμαντοι, ανύπαρκτοι, κύριε Κάνιας και Σιωδαδάνος. Και κύριοι από το Ρινιού και του Σιουδαδάνο να φέρνετε εδώ στο Κοινοβούλιο προτάσεις επικοδομητικές για λύσεις για να ανακουφιστεί ο λαός της Βενεζουέλας και τα δεινά του. Ελάτε μαζί μας να βρούμε λύσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ δεν υπάρχει λόγος. Και τι έγινε τώρα, η αντιπρόεδρος Βενεζουέλας δεν ε, πέρασε από κανένα έλεγχο διαβατηρίων, ούτε πάτησε το πόδι της στη ζώνη Σέγγεν. Και θα βοηθήσουν όλα αυτά το λαιό της Βενεζουέλας. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ να αναζητεί μια δημοκρατική λύση. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ούτε εδώ θα επιτρέψω μπλε κάρτα. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η συνάδελφος Σαράντσοβα. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται είμαι η μόνη ξένη σε αυτή τη συζήτηση, μη Ισπανή, αλλά μιλώ Ισπανικά. Σήμερα έχουμε αυτή τη συζήτηση γιατί εχθές η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπερψήφισε την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη. Και λυπάμαι που έχει γίνει η εθνική ισπανική συζήτηση όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές κυρώσεις. Και αυτό διακυβεύεται ακριβώς η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περίπτωση πλήττεται σοβαρά η αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών στη Βενεζουέλα που περιμένουν και δικαιοσύνη και στήριξη από μας. Εσείς και μάλιστα όσοι ήσασταν εδώ την περασμένη θητεία, ξέρετε ότι κάθε φορά που συζητούσαμε για τη Βενεζουέλα έλεγα το ίδιο. Επιλεκτικές κυρώσεις. Πέρασαν τρία χρόνια μέχρι να δεήσει το Συμβούλιο να κάνει το πρώτο βήμα. Οι επιλεκτικές κυρώσεις είναι ένα ειρηνικό εργαλείο πάρα πολύ ισχυρό, το ισχυρότερο που έχουμε για να πιέσουμε το καθεστώς έτσι ώστε να διαπραγματευτεί και να σταματήσει η βίαιη καταστολή του λαού της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Σαρανσοβά. Ε, θέλετε ε, ερώτηση από τον ε, συνάδελφο Καρθία Ντεμπλάνκο. Ε, δέχεστε την μπλε κάρτα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Α, τώρα ακούγεται, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, αγαπητή συνάδελφε. Εκφράζετε τη θλίψη σας ότι έχει γίνει ισπανική συζήτηση. Μα τι περιμένατε προφανές είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να γίνει η συζήτηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Ισπανική Βουλή. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Μια ομάδα, πολιτική ομάδα που δεν έχει πολιτική στέγη και ψάχνεται, προσπαθεί να δει πού θα το πάει και τι αρμοδιότητες έχει κάθε κοινοβούλιο. Δεν θεωρείτε ότι σας έχουν προδώσει οι συνάδελφοί σας ε, του κόμματος Ιουδαδάνος. Η κυρία Χαραντσοβά. Εσείς καταψηφίσατε την έρευνα στην Ισπανική Βουλή σήμερα. Και αυτό γίνεται η συζήτηση εδώ. Και όπως σας είπα, είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκές οι κυρώσεις και διακυβεύεται η ευρωπαϊκή αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χαράντσοβα. Για ένα λεπτό, ο συνάδελφος Χαβιλόπεθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έρχεται τώρα να ελέγχει τι εθνικέ κυβερνήσει. Γιατί αυτό συζητάμε εδώ. Το είπε ο Γιωσέπ Μπορέι. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια και οι κυβερνήσεις που εφαρμόζουν τις κυρώσεις. Και όχι μόνο ο ίδιος. Τις τελευταίες εβδομάδες το είπαν καμιά ντουζίνα εκπρόσωποι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εκεί υπάρχουν και εκπρόσωποι του ΕΛΚ και των φιλελευθέρων ξανά και ξανά σας τα λένε. Και σήμερα αξίζει να το επενθυμίσουμε ότι απέναντι σε αυτή τη συζήτηση τι βλέπουμε. Ότι αυτό που σας νοιάζει εσά δεν είναι η Ισπανία και καθόλου η Βενεζουέλα. Δυστυχώς φέρνετε εδώ για να κρύψετε τις δικές σας πομπές ε, στην Ισπανική Βουλή. Ε, και εμεί οι σοσιαλιστές συνεχίζουμε προσιλωμένοι υπέρ τη ε, Βενεζουέλα και δεν εκμεταλλευόμαστε πολιτικά τα δεινά του λαού της. Που εσεί το κάνετε εδώ επανελειμμένα. Ο κόσμος υποφέρει. Και αυτό δεν είναι όπλο εδώ πέρα για να το χρησιμοποιούμε και ακόμα λιγότερο για να κάνουμε εθνική πολιτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Δέχεστε ε, μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Τέρτς. Κύριε Λόπεζ, δέχεστε μπλε κάρτα. Όχι, όχι, δεν δέχεται. Ωραία, περνάμε στη διαδικασία Catch Έχω πάνω από διπλάσιους αγορητές από τη χρόνο. Θα δώσω το λόγο και σε Ισπανούς συναδέλφους, αλλά και σε μη Ισπανούς. Ο συνάδελφος ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι από τα Κανάρια, κοντά στο λαό της Βενεσουέλας γιατί έχουμε μια μεγάλη παρικία από τα Κανάρια στη Βενεζουέλα. Συμμετείχα σε όλες τις συζητήσεις και έχω ε, πει στον κύριο Μπορέλο ότι σε κάθε ολομέλεια συζητάμε τη Βενεζουέλα και υποστηρίζουμε όλα τα ψηφίσματα που ζητούν δημοκρατική αλλαγή. Τούτο εδώ δεν είναι συζήτηση ούτε για τη Βενεζουέλα, ούτε για το λαό τη, ούτε καν για την Ισπανία. Είναι μια ε, συζήτηση που έχει φέρει αντιπολίτευση κατά τη ισπανική κυβέρνηση γιατί είστε μειοψηφία στην Ισπανική Βουλή και πολλαπλασιάζονται εδώ οι συζητήσει και θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και βλάπτετε εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί τίποτα δεν βλάπτει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο η διέρεση στο εσωτερικό του και ε, προσπαθείτε εσείς να επικρίνετε την κυβέρνηση της Ισπανίας ε, με πρόφαση τα δεινά του βενεζουαλικού λαού. Μη γελιοποιήστε ε, σταματήστε πια, βοηθήστε το λαό της Βενεζουέλας και μην φέρνετε εδώ ε, αυτή τη συζήτηση που μόνο στόχο έχει να, ε, να επικρίνει την κυβέρνηση της Ισπανίας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κέλεχερ. Δεν θέλει ο κύριος Κέλεχερ. Ή απουσιάζει. Όχι, όχι, καλύφθηκε. Εντάξει. Εδώ είναι. Ε, ο συνάδελφος Φερέιρα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν υπήρχε οποιαδήποτε ανάγκη να γίνει η συζήτηση αυτή Το μόνο πράγμα που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή είναι να αναδεικνύεται το πρόσωπο, το προσωπείο του μίσου που χαρακτηρίζει την ε, ισπανική δεξιά. Αν είχαν άλλο στόχο θα υπέβαλαν ενδεχομένως κάποιους ε, αναλογικούς στόχους. Η, το ζήτημα της μη αναγνώρισης κυβέρνησης η οποία έχει εκλεγεί σε απανοτές ε, εκλογές και η υποστήριξη του αχυρανθρώπου του Τραμπ που έχει χάσει όπου και αν έχει κατέβει σε εκλογές είναι χαρακτηριστικό της στάσης των, ε, της ε, ισπανικής διεξιάς και του μίσους που την χαρακτηρίζει. Γι' αυτό και χάνεται σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ με τη συζήτηση αυτή έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι απέναντι στο πείσμα ενός παιδιού που του έχει σπάσει το παιχνίδι του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κυρία Ρέγκο, βλέπει κάποιον που έχει χάσει τις εκλογές στη χώρα του και συνεχίζει μια συζήτηση που ακόμα και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει κλείσει. Η κυβέρνησή μας κάνει μια προσπάθεια αυξάνει τον κατώτατο μισθό για να ζουν καλύτερα οι οικογένειες των εργαζομένων. Ενισχύει ε, τις ε, δημόσιες υπηρεσίες. Και εσείς εδώ και αλλού το χαβά σα. Ε, φανατικό βέτο, παρακόλληση και τα έχετε κάνει και πλακάκια με τους φίλους σας της ακροδεξιάς. Κάντε μας τη χάρη λοιπόν και ε, σταματήστε και ε, σήμερα και στο μέλλον αυτά τα καπρίτσια. Λίγο περισσότερη σοβαρότητα περιμένουμε και λίγο περισσότερη δουλειά για τα συμφέροντα του λαού μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Ντέλη έχει ω τελευταία στη διαδικασία HDI. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πραγματικά αστείο το ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε αυτέ τι διθιώτε, ανούσια ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αν γινόταν κάτι θετικό από την αντίπαλη πλευρά, πραγματικά θα τον αγνώριζα και πραγματικά θα υποστήριζα το διάλογο αν πραγματικά τον θέλανε αλλά Πώ νομίζετε ότι μπορεί να επιληθεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αυτό θα πρέπει να συζητάμε. Να συζητάμε την πραγματική κατάσταση. Ενώ αυτή τη στιγμή φαίνεται να υποστηρίζουμε έναν φανταστικό πρόεδρο, τον Γουαϊδό, ο οποίο υποστηρίζεται από τι ΗΠΑ, προσπάθησαν ουσιαστικά να κάνουν ένα πραξικόπημα στην Βενεζουέλα. Νομίζω ότι με αυτό το ζήτημα θα έπρεπε πραγματικά να ασχολούμαστε με τι πραγματικέ επιπτώσει που έχουν οι κυρώσει στο λαό τη Βενεζουέλα δυσκολίες που τους έχει προκαλέσει. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα έπρεπε να μας απασχολεί και θα έπρεπε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να δώσουμε τέλος στο εφιάλτη που ζουν οι πολίτες της Βενεζουέλα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε daily. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch και ξαναδίνουμε το λόγο στον το εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον ε, κύριο Μπορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όντως ευρωπαϊκές είναι οι κυρώσεις, αλλά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες αρμόδια για την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων αλλά και την παρακολούθησή τους είναι των κρατών μελών. Και αυτό ευρωπαϊκοί κανόνες είναι ή μήπω όχι. Για να αλλάξουν χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων. Εσείς γνωρίζετε ή θα έπρεπε να γνωρίζετε κάλλιστα ότι αυτό το θέμα του περιορισμού των ταξιδίων είναι αποφάσεις του Συμβουλίου. Άρα δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του ευρωπαϊκού νόμου. Δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι union law στα αγγλικά. Ένας πολίτης καθημερινός μπορεί να εκπλαγεί που δεν είναι η δήμον σε αυτά τα θέματα, αλλά εσείς δεν, δεν μπορείτε να εκπλήσεστε. Τι σας εκπλήσει. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου. Άρα δεν είναι κοινοτική ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενωσιακή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν έχει κανένα ρόλο στον έλεγχο της εφαρμογής. Ούτε μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάση. Εσείς είστε ευρωβουλευτές. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα γνωρίζετε. Τι σας εκπλήξει. Εμένα με εκπλήσει. Να μελετάτε λίγο περισσότερο. Δεν σας βρίσκω πολύ μελετηρούς. Απόφαση του Συμβουλίου. Συγγνώμη. Απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό το ξέρετε και το καλοξέρετε. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει ούτε να αρχίσει προσφυγή επί παραβάση. Και σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε, σας είπα, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια και θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή όλων αυτών. Άρα, είναι ένας ευρωπαϊκός κανόνας που οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και να ελέγχουν την εν λόγω εφαρμογή πάντα τα κράτη-μέλη. Πού είναι το λογικό σφάλμα σε αυτό μου το συλλογισμό. Γιατί αν δεν έχω εγώ, ε, λογικό σφάλμα το έχετε εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Επόμενο σημείο είναι δήλωση του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, είπα του εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο σχέδιο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή. Ε, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Θέλω να σας υπενθυμίσω και σε αυτή την περίπτωση, καθώς αλλάζει θέση ο Επίτροπος, ότι θα δοθεί